Przewodniczący! Dzień dobry Państwu. Καλημέρα σα. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Νούνιο Μέλο από την Πορτογαλία για μια προσωπική δήλωση. Is Mr. Mello present? Είναι παρόν ο κύριος Νούνιο Μέλο. Uh, no, he's not there at the moment. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Θα μιλήσω πολωνικά. Έχετε λάβει τα πρακτικά της ε, χθεσινής ημέρας. Υπάρχουν παρατηρήσεις για το κείμενο των πρακτικών που έχετε λάβει. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα χθεσινά πρακτικά. Και περνάμε στις ψηφοφορίες.